Dear colleagues, if you don't Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην ε, συνεδρίαση σύστασης σε σώμα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Ε, πρόσφατα ρυθμίστηκε το θέμα αυτό στον κανονισμό. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ε, συνεδρίαση σύσταση σε σώμα και επίσης ε, την εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού. Ξεκινάμε με την εκλογή του Προέδρου. Έχουμε εδώ κάποιους αναπληρωτές, κανέναν από το ΕΛΚ, από το S&D, ε, ε, ε, ο Μαντελβό θα αντικαταστήσει τον κύριο και ο Νίλ Τόρβαλς θα αντικαταστήσει τον Τόρβαλ Νίλσεν και ο Μπας Έκχουτ θα αντικαταστήσει τον κύριο Όρτασον και ο Ντέιβιτ Κόμπερν θα αντικαταστήσει η Πέτριξ Σουδόρ. Αυτοί λοιπόν είναι οι αναπληρωτές. Δεν έχει δηλώσει κανείς άλλος εξετάζουμε αν έχουμε απαρτία. Θα πρέπει να έχουμε πάνω από 16 ευρωβουλευτές. Ε, πράγματι έχουμε πάνω από 16. Ε, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει απαρτία. Ε, θα ήθελα τώρα να ακούσω τις προτάσεις για Προέδρους. Υπερβάνς Περέζ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εν ενεργεία. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να προτείνω το Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη ως πρόεδρο της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Εάν όχι, ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη ε, προτείνεται από τους σοσιαλιστές. Συμφωνείτε με την υποψηφιότητα. Παρακαλώ. ο υποψήφιος είναι κανονικό μέλος της Επιτροπής, συμφωνεί με την ε, υποψηφιότητά του και έχει υποβάλει δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία εφόσον δεν έχουν προταθεί άλλες υποψηφιότητες και δεν υπάρχει καμία ε, ε, πρόταση για μυστική ψηφοφορία. Θα γίνει η ψηφοφορία διαβοής. Ο Ρόμπερτο Γκουαλτιέρη λοιπόν εκλέγεται διαβοής και τον ε, παρακαλώ να έρθει εδώ στην θέση του. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την επανεκλογή ε, και δεσμεύομαι να εργαστώ εις όφελος ε, της, ε, των συμφερόντων της Επιτροπής αυτής με κάθε δέσμευση ούτε ώστε να συμβάλλουμε στην χάραξη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής εκπληρώνοντας και όλες τις άλλες λειτουργίες που έχει η Επιτροπή αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι λόγος για, ομιλία, για ομιλίες. Τώρα θα περάσουμε στην ε, εκλογή του πρώτου Αντιπροέδρου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν, υπάρχουν υποψηφιότητες. Κύριε Μπάλτς, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και από τη δική μου πλευρά συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας βεβαίως και εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να προτείνω τον συνάδελφο κύριο Μάρκους Φέρμπερ ως πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Αυτά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνεί ο κύριος Φέρμπερ με την υποψηφιότητά του. Ναι, φυσικά, λέει ο κύριο Φέρμπερ. Γνωρίζω ότι ο υποψήφιο είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής και έχει υποβάλει δήλωση οικονομικών ε, συμφερόντων, δεν ξέρω. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, όχι, άρα δεν υπάρχει ε, επίση και κανένα αίτημα για διεξαγωγή μυστική ψηφορία. άρα μπορεί να εκλεγεί διαβοή ο κύριος Φέρμπερ. And I invite you to join me here. Παρακαλώ να έρθετε εδώ στο Προεδρείο μαζί μου. Και τώρα θα περάσουμε στην εκλογή των άλλων λοιπόν, αντιπροέδρων. Ωστόσο, θα γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο της, τροπο, τροποποίησης του κανονισμού έχει υπάρξει μια νέα διάταξη στο άρθρο 1.2.4 το οποίο απαγορεύει την εκλογή ενός προεδρείου που να απαρτίζεται από μία, που τα μέλη του να προέρχονται από μία εθνικότητα ή να ανήκουν στο ίδιο φύλλο. Ε, θα ήθελα να ζητήσω, ζήτησα τα νόματα των υποψηφίων, αλλά φαίνεται ότι παραβιάζεται η διάταξη αυτή και προτείνω να ανασταλεί τώρα το τμήμα αυτής, ε, αυτό το τμήμα της συνεδρίασης του, της σύστασης του Προεδρείου, της εκλογής του Προεδρείου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο να λύσουμε το πρόβλημα, ούτως ώστε να συσταθεί ένα προεδρείο το οποίο να είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Θα ανασταλεί λοιπόν αυτή τη στιγμή η εκλογή των αντιπροέδρων και ζητώ από τις πολιτικές ομάδες να βρουν μια λύση το ταχύτερο δυνατό, ούτω ώστε η Επιτροπή αυτή να έχει ε, ένα πλήρες ε, προεδρείο ε, και να μπορεί να εργαστεί κανονικά. Κυρία Μπερές έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ο κανόνας 204 του νέου κανονισμού ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί προβλέπει την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και θέλει να υπάρχουν ε, βουλευτές από πολλές χώρες. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, αυτοί οι οποίοι θα εκλέγονται ε, αυτό ο οποίος θα εκλέγει δεύτερο αντιπρόεδρος είναι μέλος της ομάδας μου και θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια δέσμευση η οποία θα πρέπει να ισχύσει, να ισχύσει για το μέλλον γιατί βλέποντας την ισορροπία την οποία έχουν επιτύχει οι διάφορες πολιτικές ομάδες όσον αφορά την κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών στις διάφορες επιτροπές η δική μου ομάδα έχει το δεύτερο ρεκόρ όσον αφορά την γυναική εκπροσώπηση. Ο Χρυσούς Φίνικας βέβαια ε, πηγαίνει στους ε, πράσινους γιατί έχουν 63% γυναίκας και οι σοσιαλιστές ε, συμπεριλαμβάνομενοι στις επιτροπ... της παρουσίας ενός άνδρα έχουν υψηλό ποσοστό 80% γυναίκες και οι φιλελεύθεροι. Άρα δεν είναι δυνατόν να είναι θύμα ε, της στήριξης αυτού του κανόνα η σοσιαλιστική ομάδα. Αλλά και από αυτή την άποψη θα πρέπει να πω ότι το ECR με 12,5% γυναίκες στις θέσεις των αντιπροέδρων των επιτροπών ε, παρουσιάζει ένα έκδηλο έλλειμμα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι βέβαιος ότι οι πολιτικές ομάδες θα συμπεριλάβουν, θα λάβουν υπόψη τους αυτό το στοιχείο. Ο κ. Πάλτς, αλλά δεν πρόκειται να γίνει μια διαδικσοδική συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα κλείσει εδώ ο κατάλογος των ομιλητών, αλλά μετά θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα ρητά να χαιρετήσω εκ μέρους της ομάδας του ΕΛΚ το γεγονό ότι υποβάλλατε αυτή την πρόταση, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει εν ηρεμία να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και εγώ συμφωνώ, όπως και η Περβάνς Μπερέσε, ότι το άρθρο 204 του κανονισμού μας είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και κανονικά. Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι και για, την, ε, για το ΑΕΛΚ ότι με το ίμιση ε, ε, των θέσεων των αντιπροέδρων να έχει ήδη ε, καλυφθεί. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρότασή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την κυρία Περβάνς Μπερές. Αν ναι, η Επιτροπή κάποια ημέρα των ημερών να θεωρήσει πως η ομάδα μας είναι αρκετά καλή για να υποβάλει υποψηφιότητα για έναν αντιπρόεδρο, θα υποβάλουμε γυναίκα. Ε, Μαρίζα, quickly please. Yes, uh, quickly, just to know when do we have the election, the second... Εμείς ε, για το δεύτερο τμήμα της εκλογής, ε, τι θα, ε, θα, εντάξει, θα σας ενημερώσουμε μόλις όσο γίνεται πιο σύντομα. So we can move uh, uh, to the next point, uh, uh, elect adoption of the agenda. I ask if... ε, λοιπόν, τώρα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε αντίρρηση? ή Όχι, δεν έχετε αντίρρηση. Έχω κάποιες ανακοινώσεις εγώ. Ενημέρωση για τους συνεχιζόμενους τριμερείς. Στις 9 Ιανουαρίου έγινε, έγινε για δύο φάκελους ε, Καλύψαμε την ε, δέουσα επιμέλεια, τη διαφάνεια και τις ε, σχετικές απαιτήσει καθώς και σχετικές προσθήκες που ε, έκανε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Συμφώνησαν ότι οι περισσότερες διατάξεις για την δέουσα επιμέλεια θα εξεταστούν σε τεχνικό επίπεδο. Συμφώνησαν για τη διαφάνεια επί τη βάση τεχνικού input από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο Επόμενο τριμερής για τις 7 Φεβρουαρίου. για εις βάθος συζητήσεις θα ξεκινήσουν ίσως τότε. Σημείο 8 της ημερησίας. Ο Υπουργός έχει καταφτάσει. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα, ναι. Ήμουν ε, έτσι ταραχμένος λόγω των εκλογών. Να καλωσορίσω το φίλο και πρώην συνάδελφο Έντουαρντ Σικλούνερ που είναι πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, Υπουργός Οικονομικών, Οικονομίας της Μάλτας. Να συγχαρώ τη Μάλτα για την ανάληψη της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου για το εξάμενο αυτό. Θα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά μαζί σας ε, με θετικό πνεύμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, να βρούμε σωστές λύσεις, να φτιάξουμε σωστή νομοθεσία, καλή νομοθεσία και να ολοκληρώσουμε τους τριμερείς, ε, τουλάχιστον τους πιο σημαντικούς, όχι όλους, αλλά κάποιους όπου είναι πολύ σημαντικοί και όπου δέσμευσή μας είναι να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται περισσότερους μέσα στο δικό σας εξάμεινο. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο για τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσεις, όσοι Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, Κύριε Κουαλτιέρη, θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ καθώς και τον ε, Αντιπρόεδρο για την, εκλογή του, για την επανεκλογή για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Για μένα είναι συγκινητικό να βρίσκομαι πάλι εδώ σήμερα στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, ε, στην οποία υπηρέτησα ως Αντιπρόεδρος επί τέσσερα χρόνια. Σήμερα βέβαια βρίσκομαι εδώ με διαφορετική ιδιότητα. Εκπροσωπώ το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και θα σας παρουσιάσω τις βασικές προτεραιότητες του εξαμήνου της Προεδρίας μας. Στον τομέα Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το κάνω επειδή φαίνεται να υπάρχει μια παρεξήγηση. Υπάρχει παράδοση να παρουσιάζουν οι προεδρεύοντες του Συμβουλίου το πρόγραμμα του, της Προεδρίας στην Αρμόδια Επιτροπή. Σήμερα, λοιπόν, ε, θα παρουσιάσω τις προτεραιότητες εδώ και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι, ε, το, ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα με την ιδιότητα του Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Επιμέρους θέματα που αφορούν μεμονωμένες χώρες ε, θα πρέπει να συζητηθούν σε διαφορετικό φόρουμ στην μόνιμη επιτροπή. Χθε απάντησα, είπα ότι φυσικά είμαι στη διάθεσή τους. Και περνάμε τώρα στο πρόγραμμα της Προεδρίας. Η Μάλτα αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια χρονική στιγμή όπου η Μάλτα ε, ε, μπαίνει στο τέταρτο έτος ε, ανάκαμψης. Ωστόσο, παρά την, ε, τις θετικές εξελίξεις, η βραχυπρόθεσμη αντοχή δεν ε, σημαίνει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Μερικές φορές απογοητευόμαστε και ιδιαίτερα ε, επειδή εργαζόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης αβεβαιότητας. Κάποια από τα γεγονότα της προηγούμενης ε, χρονιάς ε, ελπίζουμε ότι θα λυθούν στην πορεία. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, η Προεδρία έχει σκοπό να αναλάβει τις ευθύνες της και θα το κάνει αυτό σε πνεύμα συνεργασίας. Είναι αλήθεια ότι η μέρος των αρμοδιοτήτων ανήκει στο Eurogroup. Αλλά και ως Προεδρία και συμμετέχοντες στην ΕΚΟΦΗΝ μας ενδιαφέρει η οικονομική ανάπτυξη. Ας ξεκινήσω όμως από τις εργασίες του Συμβουλίου στον τομέα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τον ε, Σεπτέμβριο υπέβαλε δέσμη μέτρων ε, με καινοτόμα μέτρα τα οποία εκ των οποίων κάποια ήταν αρκετά επίμαχα, αρκετοί υπουργοί θεώρησαν ότι δεν θα πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις στην οικονομική τους πολιτική. Οι συζητήσεις συνεχίζονται όσον αφορά την υιοθέτηση του, της θέσης του Συμβουλίου και κατόπιν ε, της καθοδήγησης που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο, ε, θα συμμετάσχω και εγώ στην Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Η Προεδρία προσβλέπει στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για επικαιροποίηση των ε, CSR, των κεφαλαϊκών απαιτήσεων και προσβλέπουμε στην υιοθέτησή τους μέχρι το καλοκαίρι. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές, είναι απαραίτητη η συνέχιση της εφαρμογής τους για να ξεκλειδώσουμε την παραγωγική ικανότητα των οικονομιών μας. Ε, θέλουμε επίσης ε, αυξημένη οικειοποίηση των πολιτικών της Ευρώπης ε, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει την πρόοδο. Όσον αφορά την εφαρμογή των περσινών CSR. Επίσης πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Κάτι που θυμάμαι ότι συζητούσαμε εδώ στην ΕΚΟΝ τότε που ήμουν και εγώ ε, ευρωβουλευτής. Επίσης είναι απαραίτητες αυξημένες δημόσιες επενδύσεις. Χρειάζεται όμως επίσης να είμαστε προσεκτικοί και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε συνεπή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την ε, χρήση του δημοσιονομικού χώρου και την ε, δημοσιονομική βιωσιμότητα. Κάτι που με φέρνει στην ευρωπαϊκή διάσταση, στην πολιτική ανταπόκριση στις τελευταίες προκλήσεις. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την γενική προσέγγιση πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση εν ευθέτω χρόνο. Ε, ελπίζουμε επίσης να ολοκληρωθούν εν ευθέτω χρόνο οι τριμερείς διάλογοι που ξεκίνησαν αυτόν τον μήνα. Γνωρίζουμε ότι κάποιες χώρες ε, περισσότερο από άλλες χρειάζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης ε, θεωρούμε ότι είναι δεδομένο. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως θα πραγματοποιηθεί ε, ο δεύτερος τριμερής διάλογος ε, σήμερα. Επίσης, όσον αφορά τις επενδύσεις, η Μαλτέζικη Προεδρία είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί σας πάνω στην ενδιάμεση αναθεώρηση Ε, επειδή λύγει και η θητεία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κάθε Προεδρία έχει τη δυνατότητα να οργανώσει άτυπη συνάντηση στη χώρα της και αυτό είναι μια ε, δυνατότητα που θα εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Και ε, όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, θέλουμε να ασχοληθούμε με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα εξετάσουμε και την Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, ε, θα εξετάσουμε το θέμα της φορολογικής ασφάλειας. Θέλουμε όμως να ασχοληθούμε και με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς στη Μεσόγειο που έχει να κάνει με τους οικονομικούς μετανάστες, όχι τους πρόσφυγες. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες της Βόρειας Αφρικής με ένα ε, εκτεταμένο εύση. Ενδεχομένως ε, με ένα πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενισχύσει τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, διότι αυτές αποτελούν την πύλη για τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Είναι θέμα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Χθε ε, ε, στο Παρίσι είχα συνάντηση 5 συν 5 πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη Μεσόγειο και πέντε βορειοαφρικανικές χώρες. μα ενδιαφέρει πάρα πολύ λοιπόν ε, η παράταση αυτής της εντολής ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, η ολοκλήρωσή της ε, είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης και ένα θέμα εδώ είναι το έντις. Θα πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στον επιμερισμό του κινδύνου και την μείωση του κινδύνου. Έχουν υποβληθεί διάφορες προτάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα για την μείωση του κινδύνου και παρά τις ε, τεχνικές προκλήσει και τις πολιτικές ευαισθησίε γύρω από αυτό το θέμα, η Μαλτέζικη Προεδρία θα προωθήσει τις εργασίες ε, για να ξεκαθαριστούν ε, ιδιαίτερα τα τεχνικά ζητήματα και να ολοκληρωθεί η πρόταση. Στο μεταξύ, τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην Τραπεζική Ένωση, τηρώντας τους κανόνες που έχουμε συμφωνήσει. Αυτό είναι απαραίτητο. Όσον αφορά την Ένωση Κεφαλαία Αγορών, θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Τα χαρτοφυλάκια δεν είναι πολλά στο μέτωπο αυτό, αλλά Θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή την εβδομάδα καθώς και την επόμενη όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να πετύχουμε πολιτική συμφωνία πάνω στο θέμα αυτό με το Ευρωκοινοβούλιο πριν το καλοκαίρι. Έχουμε επίσης ε, τα ε, ευρωπαϊκά, την πρόταση για τα κεφάλαια τα επενδυτικά ε, και άλλες προτάσεις. Ελπίζουμε όμως ότι θα υποβληθούν και άλλες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και στον τομέα του fintech ή του crowdfunding της ε, μαζικής χρηματοδότησης ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε νέες προτάσεις. Προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών, ε, των ε, κανονισμό για την ε, παροχή υπηρεσιών και επίσης ε, για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Προεδρία αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ισχυρές θέσεις όσον αφορά τα φορολογικά θέματα γνωρίζουμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε των θεσμικών οργάνων. Επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μα να προωθήσουμε τι εργασίε πάνω σε θέματα φορολογικά, διότι πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ορμή την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Ελπίζουμε λοιπόν τον Φεβρουάριο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. και να προχωρήσουμε στα, στις δέσμες μέτρων για, για το διπλό και τριπλό CTB. Ξέρουμε ότι οι προσπάθειες στο παρελθόν απέτυχαν. Έχει αλλάξει όμως το περιβάλλον και ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το τριπλό CTB όμως ε, παρότι θεωρείται δεύτερη φάση του θέματος αυτού, εμείς θέλουμε να θεωρήσουμε ότι αποτελεί μία ενότητα με το διπλό CTB. Κατόπιν έχουμε τη δεσμέτρων για το ΦΠΑ και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και κάτι που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας εδώ πέρα, που δεν έχει κλείσει ακόμα όμως, είναι το FTT. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για την παγκόσμια εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε την ε, ε, οικονομική και νομισματική αγορά και περιμένουμε λευκή βίβλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβληθεί σε στιγμή μεγάλης αβεβαιότητας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα περιέχει. Και Όπως είπα νωρίτερα, ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε πρόοδο. Το Συμβούλιο ε, θα εργαστεί με βάση αυτά. Ε, θα κλείσω εδώ την ομιλία μου και περιμένω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. first speaker is for the EPP Group. Thank you, Chair. Um, first of all... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Μπάλς, καταρχάς θέλω να σας ε, χαιρετήσω. Να καλωσορίσω και πάλι στην Επιτροπή μας ε, τον ε, πρώην συνάδελφο. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο θέμα του Brexit. Θέλω να θέσω αυτό το θέμα γιατί με απασχολεί. Αν η Βρετανική κυβέρνηση προχωρήσει στο Brexit, θα χρειαστεί η Προεδρία σας να ξεκινήσει τη διαδικασία. Εσείς πώς βλέπετε τη συζήτηση όσον αφορά την προετοιμασία των κατευθυντηρίων γραμμών από πλευρά της Κομισιόν. Πώς έχουν προχωρήσει οι προετοιμασίε τη ε, προεδρία σα για το συγκεκριμένο στοιχείο τη διαδικασία του Brexit και προβλέπετε διαδικασία από κάτω προ τα πάνω ή αντίστροφα. Πιστεύετε Κάποιε γενικέ δηλαδή κατευθυντήριες γραμμές ε, στην αρχή και να προχωρήσετε μετά σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις για συγκεκριμένα θέματα. Έχετε κάποια ε, σκεφτεί πώ θα προχωρήσετε. Ναι, μπορούμε να συζητήσουμε την προσέγγιση για το πώς δηλαδή θα εξετάσουμε, ε, θα, θα, θα διαπραγματευτούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς θέλουμε να είμαστε ένας έντιμος διαπραγματευτής, χωρίς να πάρουμε το μέρος κανένα. Είναι πολύ δύσκολο και στην ουσία μιλάμε στον αέρα γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 50, ε, ιδιαίτερα τώρα που το Κοινοβούλιο της Βρετανίας πρέπει να το ε, εγκρίνει το ίδιο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ε, πέρα από την προσέγγιση που έχουμε σκεφτεί, θα θέλαμε να είναι πιο κεντρικού τύπου, δηλαδή να ε, είναι σε τεχνικό επίπεδο Όσο γίνεται πιο ομαλή η διαδικασία, εάν φυσικά στην πορεία επιπλακεί, εντάξει, όλοι έχουμε τις απόψεις μας, θέλουμε να κάνουμε δηλώσεις, είτε είναι το Συμβούλιο, είτε είναι το Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε αυτό να το σταματήσουμε, αλλά εμείς θα θέλαμε να είναι πιο κεντρική η διαδικασία. και να προσπαθούμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να ηρεμούμε την κατάσταση γιατί δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να αρχίσουμε να παθιαζόμαστε και να ακολουθούμε τα άκρα και να πηγαίνουμε μάλλον στα άκρα. Είναι ένα διαζύγιο, ας γίνει όσο γίνεται πιο συνενετικό, δεν θα είναι εύκολο, εντάξει το ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα θέλαμε η διαδικασία να έχει κεντρικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ, υπερβάνω Μπερέζ. Euh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Μου κάνει... Ε, είναι σαν μεγάλη ευχαριστία που σας βλέπω εδώ και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ε, Προεδρία σας, η οποία γίνεται κάτω από μια δύσκολη συγκυρία. Ε, και αυτό είναι ένα επιπλέον λόγος για να θέσουμε κάποια δύσκολα ερωτήματα. Αναφέρετε τη σημασία της επιστροφής επενδύσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα ΕΦΣΙ είναι πολύ ουσιώδες, αλλά δεν θα είναι παρκές. Άρα ο τρόπος που θα γίνει η ολοκληρώση της οικονομικής και νομασματικής αγοράς είναι σημαντικός κρίκος. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας υπάρχουν δύο ε, συμβάντα που θα μας υποχρεώσουν να θέσουμε το ερώτημα αυτό σε σχέση με το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το πρώτο αφορά ε, το, το εργαλείο, το, άρθρο 50 και το άλλο αφορά την ε, συνθήκη της Ρώμης. Ε, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ε, της Μπρατισλάβα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ασχοληθεί με την καλή, με την εύρυθμη λειτουργία της πώς στο πλαίσιο του δικού σας χαρτοφυλακίου προτίθεστε να δράσετε, ούτε ώστε εν στην ε, σε όλα όσα θα κινητοποιηθούν εν ώψη του Brexit να μην ε, αναλωθεί όλη η ενέργεια στην υπόθεση του Brexit αλλά να δημιουργήσουμε να μετατρέψουμε το χάρτη πορείας της Ρώμης ένα, σε ένα κεντρικό εργαλείο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Γιατί η διαίρεση μεταξύ χωρών που ανήκουν στη ζώνη ευρώ και αυτές που δεν ανήκουν θεωρώ ότι είναι ένα κακό επιχείρημα για να προβάλλεται συνεχώς. Ας ξεκινήσουμε με το ε, σχέδιο Juncker. Βεβαίως όλοι εδώ είμαστε πολιτικοί και κάτι ε, το οποίο μοιάζει καλό θέλουμε να το ε, αυξήσουμε. Ε, και το σχέδιο Juncker μοιάζει θετικό. Άρα θέλουμε να, έχουμε, να το αυξήσουμε. δεν ξέρω αν μπορεί να διπλαστεί το εύση θα πρέπει να το εξετάσουμε, όπως έκανε και το ελεκτικό συνέδριο, να δούμε κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έγιναν μέχρι στιγμή σε σχέση με την αρχική μας πρόθεση. Για την προστατικότητα, για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορισμένε φορές δεν είναι δυνατόν να γίνει σε εθνικό επίπεδο ή κάτι που, έχει, που είναι, έχει ένα ιδιαίτερο ρίσκο για μια χώρα ε, ενδεχομένως ο κίνδυνος δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο Juncker. Κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί κάποια προγράμματα τα οποία βρέθηκαν, ε, ήταν καταχωνισμένα στα σιρτάρια μιας κυβέρνησης και να τα βγάλει στο τραπέζι. Γνωρίζουμε τι ευαισθησίες υπάρχουν, για παράδειγμα, σχέση με το, τους αυτοκινητοδρόμους. Ωστόσο, εγώ εκπροσωπώ το Συμβούλιο και έχω μια διαφορετική άποψη. Και νομίζω και αυτό είναι και το πνεύμα του Συμβουλίου του ΕΚΟΦΗΝ, ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα της αποτυχίας της, ε, των προβλημάτων της αγοράς. Θα ασχοληθούμε με αυτό το χαρτοφυλάκι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα αλλά νομίζω ότι είναι οι επενδύσεις υψηλότερης ποιότητας αυτές που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Όσον αφορά τους πόρους μας, ορισμένες φορές λέμε ότι μία εβδομάδα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα ε, στο πολιτικό στίβο. Τα όσα είπε ο Τραμπ σε σχέση με την κατάθμιση της Ευρώπης κλπ. Ε, ίσως ε, ενδεχομένω να μας συνασπίσουν περισσότερο. Δεν ξέρουμε ούτε καν το εφέ, το εφέ που μπορεί να έχει το αποτέλεσμα ένα tweet στις μέρες μας. Δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες εδώ, αλλά νομίζω ότι εν γέννη επιθυμούμε η Ευρώπη να πετύχει. Το θέμα είναι το πώς. Εδώ διαφωνούμε. Ορισμένοι ε, θέλουν ε, να ε, ξεκινήσουν μια κούρσα, άλλοι θέλουν να είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο διπλωματικοί και θέλουν να προσφυλθούν στους κανόνες, το πλαίσιο, δεν θέλουν να το διαρρήξουν υπάρχει ένα λεπτό όριο μεταξύ ευελιξίας και ενδεχόμενης παραβίασης των κανόνων. Ορισμένοι ε, το ερμηνεύουν σαν ευελιξία, άλλοι σαν παραβίαση κανόνων. Ε, πρόκειται λοιπόν για διαφορετικές πολιτικές ε, αποχρώσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι και αυτό ισχύει για, το, για τα διάφορα οικονομικά θέματα και για την ίδια την Τραπεζική Ένωση. Ε, η Τραπεζική Ένωση βρίσκεται σε μια πορεία δοκιμής. Ε, επιθυμούμε να πετύχουμε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να δούμε όλες τις αποχρώσεις. Όταν ξεκίνησε εδώ το σχεδιασμό του διπλού πακέτου κλπ. Δεν γνωρίζαμε τα προβλήματα που θα ανακύψουν. Ας ελπίσουμε ότι μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ευελιξία για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής ε, για το Ταμείο ΕΦΣΥ ενθουσιάστηκε με αυτά που είπατε. Πήρ Ρουχόν Λένεν από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα έγγραφα του Παναμά αποκάλυψαν ότι ο Μαλτέζος Υπουργός ε, Ενέργειας και το γραφείο του Πρωθυπουργού ε, εποφελούνταν από φορολογικό παράδεισο. Η Μάλτα μπορεί λοιπόν να ε, βρίσκεται επικεφαλής προγραμμάτων κατά της νομοποίησης παράνομων εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερη ερώτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά ωφέλη, με τα οποία προσελκύονται οι οικονομικές δραστηριότητες, είναι δυνατόν η Μάλτα να μην περνούσε την ε, δοκιμή, το τεστ ε, για τους φορολογικούς παραδείσους, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τα κριτήρια για την δίκαιη φορολογία. Και τρίτη ερώτηση. Είναι δυνατόν η Μάλτα στο μέλλον να καταλήξει στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν. Θα μπορούσα να απαντήσω και να πω ότι δεν έχω έρθει εδώ σήμερα με αυτήν την ιδιότητα, έχω έρθει ως Προεδρεύων του Συμβουλίου. Ωστόσο, ε, νομίζω ότι υπόθηκαν κάποια άδικα πράγματα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος ε, της ερώτησής σας. Ε, υπάρχουν θέματα πολιτικής διακυβέρνησης, ε, τα έγγραφα του, του Παναμά σίγουρα θα ε, οδηγήσουν στο να τεθούν τέτοια ερωτήματα και θα τα απαντήσουμε. Ωστόσο μιλάτε για άδικη φορολογία. Νομίζω όμως ότι είναι άδικο αυτό διότι δείχνει μη κατανόηση του συστήματος. Δεν πρόκειται για το κλασικό σύστημα και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ε, φορολογία και από την άλλη την ε, μυστικότητα και ε, την αποφυγή φορολογίας. Εάν κοιτάξετε την ιστοσελίδα του FIU μπορείτε να κατεβάσετε όλα αυτά τα έγγραφα που αφορούν το διάστημα πριν ε, η Μάλτα γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Μάνιβαλ ε, τα αξιολογούσε κάθε δύο-τρία χρόνια από το 1998. Ε, το τραπεζικό απόρριτο έχει αρθεί στη Μάλτα από το 1994. Αυτά νομίζω δείχνουν ότι η Μάλτα όσον αφορά τη διαφάνεια και ιδιαίτερα στην ε, ε, καταπολέμηση της ε, νομιμοποίησης παράνομων εξόδων, εσόδων όχι μόνο συμμορφώνεται απόλυτα. Θα ήθελα να σας καλέσω όμως να κατεβάσετε και τις ετήσιες εκθέσεις για να δείτε πόσα αδικήματα εντοπίζονται και καταλήγουν στο δικαστήριο. Θα δείτε με ποιες χώρες έχουμε ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες και Είμαι βέβαιος ότι αν εξετάσετε τα έγγραφα αυτά θα μιλήσετε διαφορετικά την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πίτερ Ιέσεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα δράξω την ευκαιρία αυτή να θέσω ερώτηση που ήθελα να θίξουν οι συνάδελφοι που δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε θέμα που έθιξε ο ε, Η προλαλή σας συμφωνώ ότι βρίσκεστε εδώ με την ιδιότητα του Προεδρεύοντες ε, του Συμβουλίου. Νομίζω όμως ότι η ε, Προεδρεύουσα χώρα θα πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Και όπως είπατε, η Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά θα θα κάνει μια διερευνητική επίσκεψη στην Μάλτα όσον αφορά όμως ε, το θέμα ε, της, ε, της νομοποίησης παράνομων ε, εσόδων θα συναντηθώ με δημοσιογράφο αυτή τη εβδομάδα. Αν έχετε λοιπόν θετικά νέα θα ήθελα πολύ να το ακούσω. Πάντως επί Σλοβακικής Προοδρίας οι δημοσιογράφοι δεν με ρωτούσαν τέτοια πράγματα για την Προεδρία. Κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν εδώ διότι κρίνεται σε κάποιο βαθμό η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με βάση την εικόνα της ε, χώρας της Προεδρίας. Να περάσω σε κάτι πιο θετικό. Ε, σήμερα ψηφίζουμε την οδηγία προσπέκτους για τις πληροφορίες για τα επενδυτικά μέσα και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το θέμα της τυπλοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της παρέμβασής σας. Τονίζουμε ιδιαίτερα το θέμα της ανταγωνιστικότητας για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να μειώσουμε την ανεργία. Όσον αφορά το πρώτο μέρος της παρέμβασής σας, πολύ λίγα έχω να προσθέσω. Κοιτάξτε τις πρώτες εβδομάδες ε, της Προεδρίας, δεν θα έλεγα μήνες, διότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, αλλά κοιτάξτε τις πρώτες εβδομάδες ε, πώς σκοπεύει να προχωρήσει ε, σε διάφορα θέματα και θα δείτε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Φάπιο Ντεμάζη από την ΚΟΕ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σικλούνα, είπατε ότι σήμερα βρίσκεστε εδώ με διαφορετική ιδιότητα. Κάποτε σχολίασα την φορολογία σας στην Μάλτα και μου λέτε σήμερα ότι είμαι κάποιος ε, που δεν καταλαβαίνω το φορολογικό σύστημα της Μάλτας ε, και ότι καλά θα, καλό θα ήταν να μάθω περισσότερα. Αλλά ε, είμαι βέβαιος ότι θα μας εξηγήσετε το σύστημα όταν θα βρισκόμαστε στη Μάλτα. Η Επιτροπή μας σαφώς περιμένει να μας εξηγήσετε εάν υπήρξαν ε, ποινικέ διώξεις σε σχέση με τα έγγραφα του Παναμά. σχολιάζοντας ε, την Προεδρία του Συμβουλίου, ενημερωθήκαμε ότι το Συμβούλιο αποφάσισε να μην ε, συνεργαστεί πλήρως ε, με την Επιτροπή Πάνα πρόσφατα και είναι αλήθεια αυτό και ποια είναι η προσωπική σας θέση. Μιλώ για την Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά του Κοινοβουλίου μας. Δεύτερον, επειδή ε, θα βρίσκεστε στις διαπραγματεύσεις ε, για ε, την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Ουσιαστικά έχετε οπισθοχωρήσει στην υπόσχεσή σας για τα καταπιστευματικά ταμεία. Αναφερθήκατε στο ΕΦΣΥ και την και τις προϋποθέσεις που φαίνεται να λείπουν. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας ε, επενδύσεων ε, που ε, έχει αφαιρεθεί από το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη τις κατάλληλες υποδομές. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Πολλές ερωτήσεις μου θέσατε, αλλά Όπως σας είπα, θα μπορούσα να αφήσω το θέμα αυτό για να το συζητήσουμε στη Μάλτα. Αλλά οι φορολογικές αρχές με ενημέρωσαν πριν έρθω εδώ ε, ότι όσον αφορά τα Swiss Leaks έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις έρευνες και μου έδωσαν και το ύψος του ποσού που ανέκτησαν όσον αφορά τα Panama Leaks, τις διαρροές των εγγράφων του Παναμά. Είχαμε μόλις πάνω από 100 υποθέσεις και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες εδώ και πολύ καιρό και συνεχίζονται. Όσον αφορά το θέμα των ε, δημοσίων μητρών, Ξέρω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο ακολουθεί την εξή νομική προσέγγιση. Είναι θέμα ισορροπίας. Άλλωστε, η προστασία του ιδιωτικού βίου και η προστασία των δεδομένων είναι επίσης κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, θέλουμε να υπάρχει και διαφάνεια. Δεν είναι η θέση της Μάλτας, είναι η θέση του Συμβουλίου να επιτρέψουν στις αρχές να μοιράζονται ε, δεδομένα μεταξύ τους. Οι αρχές ε, για την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα αυτή, είναι οι αρχές που έχουν σημασία στο θέμα αυτό. Υπάρχουν όμως θέματα ιδιωτικού βίου Ε, ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις. Σημαντικό είναι να μην κάνουμε κάτι που να αντίκειται ε, στην νομική τάξη και το σύνταγμα των χωρών. Έχουμε μια σχετική υπόθεση στη Γαλλία. Όσον αφορά το ευρώ υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίε. Αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρχουν τροποποίησει. σχετικά με και τον χρυσό κανόνα, θα το δούμε. Πάντως αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει κάποια ευελιξία, εξετάζονται και οι ε, υποθέσεις ε, κατά περίπτωση αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καλύτερη βάση σχετικά με την πρόταση που μου, που κάνατε. Έγινε μία ερώτηση. όχι από τη Γκουε. Ναι, ήταν ε, συνεργασία με την Επιτροπή ε, για τον Παναμά ε, και το Συμβούλιο αποφάσισε να μην συνεργαστεί. Πιστεύω πως ήταν πολύ κακή αυτή η απόφαση. Δεν είμαι ενημερός, θα ενημερωθώ και θα σας πω. Έχουμε και την συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής και θα το αναφέρω αυτό, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολ, του Πράσινη. Καλωσορίσατε. Ε, Χαίρομαι που σας βλέπω και άμεσα και όχι μόνο μέσω του τύπου της Μάλτας. Ε, στην εφημερίδα Independent της Μάλτας ε, σας ανέφεραν όσον αφορά τους στόχους ε, ε, για τη φορολογία για την προεδρία της Μάλτας. Είπατε λέει ότι η Μάλτα δεν αισθάνεται ε, άσχημα που χρησιμοποιεί τη φορολογία ως μέσο ανταγωνισμού όπως και τους μισθούς και όσον αφορά τη φορολογία κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίζει για τον εαυτό του. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τη θέση που έχουμε ακολουθήσει εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο όπου διαρκώς λέμε πως χρειάζεται κοινό πλαίσιο και για την ε, φορολογία. Η δική σας φορολογική πολιτική έχει ένα συγκεκριμένο στόχο να ε, καλέσει να προσελκύσει τις εταιρείες μέσω μιας μείωσης των φόρων ε, που τους επιβάλλεται. Μείον 5%. Αυτό οδηγεί σε μια κακή φήμη για παράδεισο φορολογικό. Αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Δεν βλέπω διαφορά ανάμεσα στο Λουξεμβούργο και τη Μάλτα, όπου το Λουξεμβούργο όταν είχε την Προεδρία έχει βάλει στο πρόγραμμα της Προεδρίας τα φορολογικά θέματα στην πρώτη θέση. Ε, σε εσά ε, ούτε καν υπάρχει το θέμα. Εσείς είπατε εντάξει ότι θα ασχοληθείτε με τη CCCTB, αλλά ε, παρότι η Κομισιόν έκανε πρόταση στις 25 ε, Οκτωβρίου, η πρώτη τεχνική φύση συνεδρίαση του Συμβούλιο έχει οριστεί μόνο για τις 16 Φεβρουαρίου. Οπότε Κοιτάξτε, προχωρήστε τα φορολογικά θέματα, ακόμα και αν δεν είναι στις, στο πρόγραμμά σας, αλλά και κοιτάξτε να συνεργαστείτε και με την Επιτροπή Πάναμα, συμπεριλαμβανόμενη της έκθεσης ε, και που μέχρι στιγμής ε, δεν έχει δημοσιευθεί. Ο κύριος ο κύριος Μάνφρον Γκάλ έχει παραιτηθεί από τη θέση του. Παρακαλώ λοιπόν να υποβάλλετε αυτό το έγγραφο και στο μαλτέζικο τύπο και σε εμά ο Υπουργό. Φοβούμαι πως δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ, γιατί αυτό που περιγράφεται είναι κομμάτι του συστήματος όπου η Κομισιόν και η, Επιτροπή, η αρμόδια για την Επιτροπή Ανταγωνισμού ε, το εξολόγησαν και εγκρίθηκε το σχέδιό μας αφού ζητήθηκαν κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν. Κάποιες εταιρείες ε, ε, αφαιρέθηκαν και εσείς επίσης. Για το σύστημά μας λοιπόν λειτουργεί και όπως οποιοδήποτε άλλο φορολογικό καθεστώς στην πράξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον. Εξαρτάται από τους ε, άμεσα ενδιαφερόμενους για το πόσο ε, ε, μπορεί κανείς να το εκμεταλλευτεί. Τώρα αν είναι ευάλωτο είναι το ίδιο ευάλωτο με άλλα συστήματα. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη διπλή μη φορολόγηση και την φοροαποφυγή. Μάλτα θα συνυπογράψει την πολυμερή συνθήκη συμφωνία του ΟΣΑ και θα, θα τηρήσουμε τις συστάσεις ΠΕΠΣ. Είναι πραγματικά καρικατούρα του να ακολουθείτε τις τίτλους, τι είπα, τι φάνηκε στις εφημερίδες κτλ. Τι λέτε για το 5% φορολογία. Όχι, είναι λάθος τότε δημοσία πρέπει να το διορθώσετε και να μας πείτε τι δεν στέκει από όλα αυτά. Ναι, αυτή η αποζημίωση ξαναφορολογείται, η επιστροφή μάλλον ξαναφορολογείται. Είναι λάθος αυτά που μου λέτε. Ευχαριστώ. Μάρκο Τζάνι, ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία ε, στον ε, Πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ για το επόμενο εξάμεινο, γιατί πιστεύω πως η κυβέρνηση της Μάλτας ε, θα πρέπει να διαχειριστεί την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια φάση πολύ δύσκολη και πολύ προβληματική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Κίνδυνοι πολιτική και οικονομική τους επόμενους μήνες για μια πιθανή κρίση με την έξοδο κάποιων μελών της Ευρωζώνης. Σήμερα αυτός ο κίνδυνος είναι πλέον αποδεκτός και από σχολιαστές με κύρος και μάλιστα ε, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας πριν από λίγες μέρες μόλις δέχτηκε την πιθανότητα μια χώρα να μπορεί να φύγει από την Ευρωζώνη. Περάσαμε από το whatever it takes του 2012 στην πιθανότητα ξόδου υπό όρους το 2017. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι σε αυτή την φάση. Η Μαλτέζικη Προεδρία στο εσωτερικό του Συμβουλίου και στο κυρίως στο εσωτερικό του ΕΚΟΦΗΝ σκοπεύει να θέσει αυτό το θέμα επιτάπητος ώστε να προκληθεί συζήτηση ανάμεσα στα κρατημέλη και μάλιστα με την συγκεκριμένη δυνατότητα κρίσης της Ευρωζώνης και κάποιες χώρας να βγει, να φτιάξετε κάποιο σχέδιο, προ, προ, προβλέψετε τι θα συμβεί αν όντω γίνει κάτι τέτοιο. Μελετάτε τι θα κάνετε. Θα φτιάξετε μηχανισμούς για να χειριστείτε μια κατάσταση που είναι συγκεκριμένη και που μπορεί να είναι πολύ προβληματική ή όπως συχνά έχετε αποαντήσει στο παρελθόν κατά τη γνώμη μου όχι με πολύ έξυπνο τρόπο δεν εξετάζετε αυτή την επιλογή και δεν εργάζεστε για ένα πλάνο B όπως λέμε ένα ε, πλάνο αντιμετώπισης μιας τέτοιας περίπτωσης σκοπεύετε να κάνετε μια επικοδομητική συζήτηση για ένα γεγονός, για, κάτι μάλλον που μπορεί πιθανότατα να συμβεί στους, επόμενου ε, στους επόμενους μήνες του 2017. Well, the Κοιτάξτε, το ECOFIN συναποτελείται από τους υπουργούς των 28 κυβερνήσεων. και όπως, όπως οποιαδήποτε κυβέρνηση και ή υπουργό δεν μπορεί να είναι ε, παρά σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τούτο λεχθέντος αυτό που θα θέλαμε είναι να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό στο άτυπο Εκοφίν θα θέσουμε το, εκο το λευκό βιβλίο ως ένα από τα τέσσερα ζητήματα που θα αποτελέσουν τη, τη βάση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Επίσης, πιο, σημαντικό είναι το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά ζητήματα. Υπάρχει όντως μεγάλη ανησυχία στο εκλογικό, που επικρατεί στο εκλογικό σώμα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και αλλού. Και φόβος. Φόβος για τη μετανάστευση, την τρομοκρατία και τη φτώχεια. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν αυτά τα θέματα μπορούμε να καθησυχάσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Αντί να αρχίζουμε να ετοιμάζουμε δεύτερο και τρίτο σχέδιο και δεν θέλω με αυτό να ελαχιστοποιήσω την σημασία του Λευκού Βιβλίου που θα έρθει μετά από την ε, συνεδρίαση της Ρώμης. Πάντως ε, πιστεύω πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Αυτό είναι ο ρόλος μας στο ΕΚΟΦΗΝ και ε, ο ρόλος μας εδώ στο, εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να μειώσουμε την αβεβαιότητα, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, να εξετάσουμε τα θέματα της μετανάστευσης και πολύ θα ήθελα εδώ να κάνω διάκριση ανάμεσα στους μετανάστες και τους οικονομικούς μετανάστες γιατί οι πρόσφυγες είναι προϊόν πολέμου, ενώ οικονομική μετανάστευση είναι προϊόν της ανισορροπίας ανάμεσα στις πλούσιες και τις στοχές χώρες. Μια ανισορροπία που θα πρέπει να την μειώσουμε γιατί αλλιώς η οικονομική μετανάστευση θα συνεχίζεται στο δυνικές. Plan B σημαίνει την αντιμετώπιση της, πιθανότητα εξόδου μιας χώρας από το ευρώ δεν πρέπει να είστε έτοιμοι. Ναι, η Κομισιόν θα πρέπει να μας ετοιμάσει αυτό το λευκό βιβλίο για το μέλλον της ε, Ένωσης. Ε, φαντάζομαι και ελπίζω ότι ε, τόσο ότι στο ΕΚΟΦΗΝ θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα και πώς θα ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Η πλατιά πλειοψηφία του Κοινοβουλίου συμμερίζεται αυτή την άποψη. Uh, κύριε Σκόμπορν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε Μαλτέζους, έχουν μακρά σύνδεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα μας ε, βοηθήσουν με την δημοκρατικά αποφασισμένη έξοδο. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει ειρηνικά η έξοδος. Θέλουμε να συνεργαστούμε βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουμε να συμβεί κάποια καταστροφή όλεθρος. Ε, και νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε. Μότο, ότι αναφέρατε ε, ε επενδύσει σύμφωνα με το σχέδιο Juncker. Εγώ μιλάω από μια φιλελεύθερη άποψη. Θεωρώ ότι το σχέδιο Juncker δεν είναι καλή ιδέα πιστεύω ότι οι κυβερνήσει δεν δημιουργούν θέσει απασχόληση, επιχειρήσει δημιουργούν θέσει απασχόληση. Και οι επιχειρήσεις ε, ε, ε, επιχειρηματίες δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και νομίζω ότι το σχέδιο Juncker πραγματικά είναι σφαλμένο. Όσον αφορά τα ασφαλιστικά, τα σταξιδιωτικά ταμεία, τα οποία πρόκειται να κάνουν επενδύσεις, ε, δεν ξέρω. Θα ήθελα η Μάλτα να ασχοληθεί με το θέμα του ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επιθυμούμε μια σταθερή Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι σημαντικός για μας και θεωρούμε ότι η Μάλτα συμφωνεί με αυτή την ιδέα και θα θέλαμε να σας δούμε να προωθήσετε αυτή την ιδέα στην, στο ΕΚΟΦΗΝ γιατί μόνο έτσι θα πάρετε τα χρήματά σας, θα, θα κερδίσετε τα χρήματά σας ε, που έχετε επενδύσει. Ε, Ε, δεν νομίζω ότι όλοι στην Ευρώπη συμμερίζονται την ιδέα της, ε, του να επενδύονται τα χρήματα ε, οπουδήποτε. Όσον αφορά το σχέδιο Juncker, το, Juncker, το σχέδιο Juncker είναι ένα κουτί το οποίο μπορούμε να το γεμίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Ε, νομίζω βασική ιδέα ήταν οι ιδιωτικέ επενδύσεις που είπαμε ότι θέλουμε να το, τις παρακολουθήσουμε και να δούμε τι ποιότητα έχει. Δεν πρόκειται για τις ε, δημόσιες ε, επενδύσεις εδώ, αλλά για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το θέμα είναι λοιπόν τι μπορούμε να πάρουμε. Βεβαίως ε, υπάρχει ένα θέμα αποτυχίας της αγοράς τομείς όπου ο κίνδυνος για τους ιδιωτικούς επενδυτές είναι υπερβολικά υψηλός. Και εδώ το δημόσιο έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο. Κατά τα άλλα, συμφωνώ ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί ε, είναι τα χρήματα κάποιων άλλων, οι οποίοι ε, βεβαίως τα διακινδυνεύουν και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να είναι ε, καλές οι επενδύσεις τους. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο Juncker, εγώ δεν θέλω να το καταδικάσω, ούτε να το επενέσω, αλλά θα πρέπει να το δούμε έτσι όπως είναι. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο B, ε, τι γίνεται με το σχέδιο B, αν ε, ε, κάποια άλλη χώρα θέλει να φύγει. Νομίζω ότι είναι προς συμφέρον όλων, ακόμα και αν εμείς δεν συμμετέχουμε, δεν είμαστε στην ζώνη ευρώ, παρόλα αυτά δεν θέλουμε η έξοδός μας να σηματοδοτήσει μια καταστροφή. Ο Γκούναρ Χόκμαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπαν ε, όλοι, καλωσορίσατε. Έχω μια σκέψη σε σχέση με τα όσα είπατε στην πρώτη σας παρέμβαση. Εν σχέση, πώς να δούμε για τους κανόνες για το σύμφωνο σταθερότητας. Εάν ε, δεν απατώμε, το ένα άλλο πράγμα είναι η παραβίαση και άλλο η ευελιξία σε σχέση με τους κανόνες. Το ερώτημα είναι γιατί έχουμε κανόνες, για να υπάρχει μεγαλύτερη εξοπιστία. Και αν ε, η Προεδρία του Συμβουλίου λέει ότι μπορεί να κάμψει, να λυγίσει τους κανόνες ε, χάρη μιας ευελιξίας, αυτό με ανησυχεί. Εάν δούμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ιδιαίτερα βραδία. Ε, η ενιαία νομισματική πολιτική δεν θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Γνωρίζουμε ότι η μεγέθυνση που έχουμε είναι πολύ άνισα καταναμημένη. Σε ορισμένες χώρες είναι υψηλή, η οικονομική ανάπτυξη, σε άλλες είναι χαμηλή. Ε, Άρα λοιπόν ορισμένες φορές ε, έχουμε σφαλμένη εικόνα από κάποια στοιχεία και οι χώρες μέλη έκαναν προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν ε, την οικονομία τους ε, σεβόμενες τους κανόνες. Αυτό το έκαναν μερικές χώρες. Άλλες κάμπτουν τους κανόνες χάρη της ευελιξίας και βλέπουμε ότι τα ελλείμματα ε, δεν ε, υποβοήθησαν την ε, ανάπτυξη, αντιθέτως επιδίνωσαν την κατάσταση. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τι γίνεται με αυτή την ευελιξία, κατά πόσο προτίθεστε να κατοχυρώσετε ως Προεδρία το σεβασμό και την τήρηση των κανόνων. Νομίζω ότι ίσως υπήρξε μια έλλειψη σαφήνειας από τη δική μου πλευρά. Εγώ δεν θεώρησα ότι θα πρέπει να παραβιάσουμε τους ε, κανόνες. Είμαι υπέρ της στήρησης των κανόνων εντός του ισχυρήνους πλαισίου. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι αν μελλοντικά κάποιος ε, θα πρέπει να σκεφτεί όλα τα σενάρια και να έχει κάποια ευελιξία η οποία βεβαίω θα πρέπει να συμφωνηθεί. Ε, ποιο είναι το περιθώριο της ευελιξία. Είναι σαν μια διακύμανση, είναι σαν ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη ε, στην περίπτωση αυτή. Αυτό ε, θέτει τα όρια της ευελιξία. Αλλά βεβαίω είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν κάποιες αποφάσει στο ΕΚΟΦΗΝ όταν πρόκειται για πακέτα για δομές που έχουμε επεξεργαστεί, αλλά αφήνοντας ε, έξω ορισμένες ε, ε, αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει, αν μια χώρα ζητήσει κάποια ευελιξία, αυτό είναι σημαντικό. Όταν φτιάξαμε αυτά τα εργαλεία, 2-pack, 4-pack κλπ, θα μπορούσαμε να έχουμε συμπεριλάβει στο σύστημα, εντάξει μέσα στο σύστημα, κάποιο περιθώριο ευελιξίας. Αυτό εννοούσα. Δεν εννοούσα μια παράκαμψη, μια ε, ε των ε, κανόνων. Ε, απλώς είπα ότι υπάρχει και ένα ζήτημα ερμηνείας εδώ και ε, είναι δύσκολες αποφάσεις, ε, ιδιαίτερα για χώρες που είναι κρίσιμη η κατάστασή τους σε συνάρτηση πάντα με την πολιτική σταθερότητα. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε είναι οι μεγάλες χώρες να την χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Αλλά βεβαίως αυτό είναι ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Αλλά πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει μια εύκολη απάντηση εδώ, γιατί από τη μία πλευρά όλοι επιθυμούμε να τηρήσουμε το πλαίσιο και όταν το φτιάξαμε, είπαμε, είδατε τι έγινε στο παρελθόν, δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι θεμητό να υπάρχουν κάποια δισταγμοί. Το ερώτημά μου είναι πώς θα αντιδράσετε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Συμφωνώ ότι πολλά πράγματα είναι δύσκολα, δυσεπίλητα. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσετε εσείς όσον αφορά τους κανόνες. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε εντός των κανόνα. Αυτή είναι η απάντησή μου εν συντομία. Σας ευχαριστώ και γνωρίζουμε ότι ε, και αυτό είναι μέσα στους κανόνες. Ο κύριος Χακμακή είναι διατησμένος να ανοίξω οποιαδήποτε συζήτηση. Ε, νομίζω ότι έλειξε ο χρόνος του νέα αλλά του Προέδρου, απαντάει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος έχει περισσότερα προνόμια. καλώ ορίσατε στην Επιτροπή σα αυτήν, την οποία γνωρίζετε καλά. Θα ήθελα πολύ να παραμείνω εντό του θέματο αυτού ε, σχετικά με την ε, παραβίαση και τήρηση των κανόνων. Ε, πρόβλημα στην Ευρωζώνη παραμένει το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. χαμηλά επίπεδα ε, δημοσίων επενδύσεων ε, σημαίνει και λιγότερες ε, ιδιωτικές δεσμεύσεις. Και το σχέδιο Juncker προσπάθησε να λύσει το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν αρκεί καθόλου. Και αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες θυσιάζονται για πολιτικούς αλλά και όχι μόνο λόγους. Εσείς πώς θα βλέπατε τη μείωση του χρυσού κανόνα που θα επιτρέψει οι καθαρές δημόσιες επενδύσεις ε, να μην ε, συνυπολογίζονται ε, και υπάρχει μεγάλη πολιτική αντίθεση. Πιστεύετε όμως ότι από τεχνικής άποψης αυτό είναι δυνατό να γίνει χωρίς να διακυβεύονται τα κριτήρια σταθερότητας. Um, Όσον αφορά τις ιδιωτικές ε, και δημόσιες επενδύσεις, ε, οι δημόσιες είναι συλλογικές και θα θέλαμε ε, όπου είναι δυνατόν να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες σε περίπτωση που από τη γάλλη αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε την ποιότητα και όχι μόνο την ποσότητα των δημοσίων επενδύσεων. Όσον αφορά το χρυσό κανόνα, ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ ακολουθώ την ε, διαδικασία που θα πρέπει και θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό στο συμφωνημένο πλαίσιο. Έχουμε το EFC. Έχουμε μια σειρά αποδομές γύρω από αυτήν τη διαδικασία. Ό,τι και να γίνει δεν μπορούμε απλά να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πανάρχομαι έτσι στις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Χακμάρκ. Ε, πρέπει να ε, ενεργήσουμε εντός του συμφωνημένου πλαισίου, αλλά αυτό βέβαια δεν αποκλείεται το να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έχετε μια δεύτερη ερώτηση, έχετε χρόνο. Δεν συνειδητοποιείτε όμως ότι ο τρόπος που χειριζόμαστε τις επενδύσεις ε, στον δημόσιο προϋπολογισμό ε, τηρούμε τον, ε, αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο τις επενδύσεις με τις δαπάνες. Έτσι λοιπόν ο κάθε υπουργός Οικονομικών έχει κίνητρο να μειώσει τις δαπάνες για να τηρήσει το χρυσό κανόνα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δεν το βλέπετε. Όπως σας είπα, η προσωπική μου γνώμη είναι άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι ε, είναι εντολή των ε, κυβερνήσεων ε, και των υπουργών να συζητήσουν το θέμα αυτό. Αναθεωρούμε αυτή τη στιγμή τους κανόνες Στην ΕΚΟΦΗΝ, στο Άμστερνταμ για παράδειγμα, συζητήσαμε αν θα πρέπει να ε, ε, αλλάξουμε τον κανόνα, αντί για κανόνα περιελήμματος, να έχουμε ε, κανόνα περί δαπανών. Δεν μας εμποδίζει τίποτα να συμφωνήσουμε νέους κανόνες, όπως θα ήταν αυτός. Δεν είναι αυτή η δική μου άποψη, αλλά κατά την αναθεώρηση των κανόνων αυτών, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τον κανόνα περί χρέους και τον κανόνα περί ελλείμματος. Τίποτα δεν μας εμποδίζει κατά την αναθεώρηση αυτή να εξετάσουμε και τη δική σας πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τεχνικής πλευράς υπάρχει ένας ε, κανόνας ε, για τις επενδύσεις, αλλά είναι πολύ περιορισμένος. Υπάρχει όμως. Ο Βέρνερ Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ως Υπουργό Οικονομικών ε, της Μάλτας είσαστε διατηθειμένος να συνεργαστείτε στενά με το Κοινοβούλιο. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ε, η ε, Μαλτέζικη κυβέρνηση ήθελε να δημοσιεύσει τις ε, φορολογικές ε, συμβάσεις. Ε, πέρσι το αυτό, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Η κυβέρνηση τι θα κάνει για την φοροαποφυγή. Ε, χθες είχαμε ακρόαση κατά την οποία ένας από τους καθηγητές είπε ότι ο διαμεσολαβητής Ε, θέλει να παρακάμψει τους το πνεύμα των φορολογικών κανόνων, ε, όχι όμως το γράμμα. Είναι λοιπόν δύσκολο το θέμα αυτό. Αύριο έχουμε προβλέψει κοινή συνεδρίαση της ΕΚΟΝ και της ε, ΠΑΝΑ, της Επιτροπής για τα έγγραφα του Παναμά αλλά αναβλήθηκε αυτό διότι είπαν ότι δεν ε, έχουν έτοιμα τα έγγραφα, το οποίο δεν είναι αλήθεια και ότι θα πρέπει να βρουν άλλη στιγμή για τις συζητήσεις. Ε, ερώτηση λοιπόν, τι θα κάνετε για να πετύχετε καλύτερη συνεργασία ε, με το Κοινοβούλιο πάνω στα θέματα αυτά. Είσαστε υπέρ απεριόριστης πρόσβασης στα έγγραφα ή όπως προκύπτει από τα πρακτικά θα ακολουθήσετε την ε, θέση του Λουξεμβούργου ότι θα πρέπει ε, να ε, ενεργήσετε συγκρατημένα και να μην προσεγγίσετε τη θέση του Κοινοβουλίου. Από ό,τι γνωρίζω δεν θέλετε να επιδεινώσετε την ε, συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως να αυξήσετε την πίεση στα άλλα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα και να μην ε, γίνουμε θέαμα στο κοινό. Θα ξεκινήσουμε από το θέμα των tax rulings, των φορολογικών αποφάσεων και της Μάλτας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από κάθε κράτος μέλος τις συμβάσεις αυτές ε, και η Μάλτα απάντησε ότι δεν έχει τέτοιο σύστημα. Υπάρχει ισότητα για όλους, ε, δεν γίνονται διακρίσεις. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, δεν έχουμε τέτοιες φορολογικές αποφάσεις, tax rulings. Όπως γνωρίζετε, η φορολογία συνεχίζει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η ΕΚΟΦΗΝ, αλλά το τι γίνεται εντός των κρατών μελών. Η Επιτροπή Πάνα, όταν καλεί κυβερνήσεις να συνεργαστούν ε, με την Εξεταστική Επιτροπή, εναπόκειται στις κυβερνήσεις να απαντήσουν στην πρόσκληση. Στην δική μας περίπτωση, επιλέξατε να προχωρήσετε ακόμα πιο πέρα, να επισκεφτείτε τη χώρα μας και να ζητήσετε από ε, ε, στελέχη συμπεριλαμβανομένου εμού να συνεργαστούμε με την Επιτροπή. Ωστόσο, και ελπίζω να μην κάνω λάθος, ε, πιστεύω ότι το θέμα του χειρισμού των εγγράφων δεν συζητήθηκε καθόλου στην ΕΚΟΦΗΝ αφέθηκε στις κυβερνήσεις να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεργαστούν ή όχι. Εναπόκειται σε αυτές να αναλάβουν ευθύνη για τις δράσεις τους. Ε, σχετικά με τα έγγραφα στα οποία αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, δεν αμφισβητώ την ε, βούλησή σας να συνεργαστείτε, αλλά από, το, τα πρακτικά προκύπτει ότι σε αντίθεση με τις ε, περισσότερες χώρες, ε, οι κάτω χώρες θέλησαν να συνεργαστούν με το με το Κοινοβούλιο, τα πρακτικά ε, καταλήγουν ε, ότι δεν είναι δυνατόν η αύξηση της συνεργασίας. Θα πρέπει εσείς λοιπόν να φροντίσετε οι άλλοι Υπουργοί Οικονομικών και οι άλλες κυβερνήσεις να συνεργαστούν καλύτερα από ό,τι μέχρι τώρα, διότι έχουμε σχετικά, λάβει σχετικά λίγα έγγραφα, ε, μην σας πω και κανένα έγγραφο. Thank Σας ευχαριστώ, το σημειώνω. Ευχαριστώ κύριος Μπούλμαν. Uh, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να σας καλωσορίσω. Χαίρομαι πολύ που σας ε, βλέπω. Έχουμε αυτήν την ε, φορολογική πολιτική εντός του ε, Συμβουλίου. Γιατί να μην κάνουμε το εξής. Η ε, ε, ο Επίτροπος είναι μάλλον υπέρ του να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο για να αξιολογηθεί η ομαδοποιημένη στα, στάση του της Ένωσης. Εμείς γιατί να μην αξιολογήσουμε το κόστος του να μην το έχουμε αυτό. Τις επιπτώσεις για την ενιαία αγορά, ε, θα μπορούσαμε να θαρρύνουμε λοιπόν την Κομισιόν να κάνει αυτή την εξέταση ώστε τελικά να κάνουμε μια πιο λογική συζήτηση για όλα αυτά. Έπειτα εκτιμώ το γεγονός ότι αναφέρθηκατε όχι μόνο στο δεδομένο πλαίσιο αλλά και στη διάσταση της οικονομικής μετανάστευσης και ο Τζοζέφα Μουσκάτ, ο Πρωθυπουργό σα ήδη αναφέρθηκε σε αυτό στην Ολομέλεια. Πολύ υπεύθυνη αυτή η στάση, αλλά πρέπει επίσης να αναφέρω, επειδή είμαι συνεισηγητής σε αυτή την υπόθεση, Μέσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, εντοπίζουμε ένα είδος ε, τεχνοκρατικής, γραφειοκρατικής ε, λειτουργίας και άρα το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει το μηχανισμό. Εσείς μπορείτε να καλέσετε τους συναδέλφους σας ώστε να εξετάσουν πιο προσεκτικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, όταν πρόκειται για τις διαστάσεις του ΕΦΣΙ ή για το επόμενο ΕΦΣΙ 2 και επίσης να μας πείτε τις ιδέες για το χρήση του ίδιου τύπου μέσου για τον διάλογο μεταξύ Βορρά και Νότου. Εγώ πολύ θα εκτιμούσα να κάνετε μια, ένα τέτοιο διάλογο ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. separate meeting with the social. Yeah. Well, I'm being informed that we have both a macroeconomic dialogue, but also regarding the fiscal policy stance. Για την θέση την, της, για την φορολογική πολιτική, την οικονομική πολιτική, η Προεδρία πρέπει να σας πω ότι Κάπως εκνευρίστηκαν διάφορα κράτη. Η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση της ε, οικονομικής ε, ε, θέσης και στάσης. Γιατί ήταν κάτι το οποίο είχαν συμφωνήσει πριν και κάπως εξεπλάγησαν όταν συνέβη είναι ένας τομέας ε, φεός Σίγουρα θέλουμε πρόοδο εδώ. Ο συντονισμός είναι ούτως ή άλλως ο στόχος, ο τελικός στόχος και πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα τον επιτύχουμε. Σε σχέση με την, ε, με την ε, ΤΕΠ, αυτή παρακολουθεί τις, συν, συνεδριάσεις ε, του ΕΚΟΦΗΝ πρέπει να πω ότι τα θέματα τα οποία αναφέρατε δεν έχουν συζητηθεί στο παρελθόν, από όσο θυμάμαι. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα κρατημέλη και την ε, ε, ΕΤΕΠ. Ίσως θα μπορούσατε κάπως να διευκρινίσετε τι εννοείτε. Ναι, ευχαρίστως. Ποιος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο Τη ΤΕΠΕ, τα κρατημέλη. Άρα τα κρατημέλη είναι υπεύθυνα για την πολιτική που ακολουθείτε τελικά. Και αν έχουμε μια εγγύηση από το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που δίδεται στην, στην ΕΤΕΠ ώστε να διευρύνει όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των επενδύσεων, τότε τα χρήματα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όχι για να μειωθούν οι ε, τακτικές ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες, ε, γιατί τότε έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλω να καλέσετε τα κατημέλη σε πλήρη συζήτηση, full συζήτηση, γιατί δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ένα μηχανισμό, ενώ στο, στη λειτουργία, στην εκτέλεση, λειτουργούμε με απρόβλεπτο τρόπο, γιατί αυτό έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά και αυτό δεν μπορεί να το επιτρέψει το Κοινοβούλιο. Ίσως να σας απογοητεύσω σήμερα, αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σημειώσω το αίτημά σας και να το λάβω σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ κύριο Σκάζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Σικλούνα. Μιλάμε πολύ για την ε, νομοθεσία κατά του ξεπλήματος χρήματος. Εσείς είστε υπεύθυνο για την, ε, ε, το γραφείο πληροφοριών της υπηρεσίες για κατά του οικονομικού εγκλήματος. Για τα έγγραφα του Παναμά, πότε θα δημοσιεύσετε αυτά τα έγγραφα, πότε θα επιλέξετε έναν νέο διευθυντή αντί για τον κύριο Γκόλτες που αναμεγνύεται σε αυτά τα σκάνδαλα και έπειτα η, διεθνής, ε, η, Ένωση Transparency International λέει ότι η Μάλτα δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Κάθε θεσμικό όργανο, το FIIU, όπως και όλα τα θεσμικά όργανα, διέπονται από την νομοθεσία και λειτουργούν με ανεξαρτησία και αυτονομία. Επίσης, αυτό που μπορούν να αποκαλύψουν ή όχι ως πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένα. Τώρα, για τον ε, διευθυντή στον οποίο αναφέρεστε, εκείνος ε, ε, έπρεπε να συντάσει αναφορές ε, με πιο βρύς όρους. Εγώ τον ενθάρρυνα σε αυτό, αλλά ποτέ δεν συζητήσαμε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ε, ποτέ δεν συζητήσαμε για μεμονωμένες εκθέσεις και θα ήταν παράνομο να κάνει ο ίδιος κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος αυτού του θεσμού της Μόλτας είναι της Μάλτας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, ενώ ο αναπληρωματικός πρόεδρος ε, προέρχεται από την υπηρεσία ελέγχου, οικονομικού ελέγχου της Μάλτας προσωπικότητα με μέγα κύρος και μάλιστα τα, καθήκο, τα προσόντα του είναι τέτοια ώστε ορίστηκε να κάνει αξιολόγηση για όλες τις ε, χώρες. Έχει μέγα κύρος, ε, και χέρι εκτιμήσεως δεν μπορώ παρά να, να βρω καλύτερα ε, ανθρώπους για να εμπιστευτώ αυτό το θεσμό. Το Dr. Μπάρτος που είναι από την ε, συγκεκριμένη υπηρεσία και τώρα επαναδιορίζεται το ίδιο συμβούλιο. Οπότε θα αγκατασταθούν, θα αναλάβουν ε, τα καθήκοντά τους. Επίσης με ενημέρωσαν ότι ότι οι συνεντεύξεις για να βρεθεί ένας ε, άνθρωπος για να αναλάβει την, ε, τη θέση που κερνούνται ε, ήταν πολύ μακρές και ότι τελικά κατάφεραν να βρουν τον, το λόγο άτομο και ότι η θα διεκπαιρωθεί η διαδικασία και θα οριστεί ε, λόγω άνθρωπος στο Συμβούλιο. Πάντως δεν έλαβα εγώ εκθέσεις για συγκεκριμένες υποθέσεις και θα ήταν παράνομο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτόνομοι και έχουν δεχτεί και να ε, μας συναντήσουν και να εξηγήσουν τη θέση τους. Και όπως είπα, η ετήσια έκθεση που εκδίδεται κάθε χρόνο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σε σχέση με τα κράτη-μέλη με τα οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, είτε είναι ας πούμε, με το Ηνωμένο Βασίλειο 35 υποθέσεις, με την Ιταλία 46, η Γαλλία 10 υποθέσεις κτλ. λοιπά Η Ελβετία 20 υποθέσεις, όπου δηλαδή συνεργάζονται με τις αρχές άλλων χωρών. Ε, πάρα πολύ σοβαρός ε, θεσμός. Είναι ατυχές όπως είπε και ο κύριος Κάζα, Είναι ατυχές που παρετήθηκε ο μέχρι τώρα διευθυντής και άλλος άνθρωπος θα αναλάβει τα ενία. Πάντως παρακαλώ να μην κρίνετε ε, τους θεσμούς, ε, να δείτε το πρόγραμμα εργασίας. Ε, θα πρέπει να δούμε αν, έχουμε το κατάλληλο σύστημα, αν καλύπτουμε κάθε είδους εγκλήματα και έπειτα τα παραπτώματα και υποθέσεις στο δικαστήριο αφορούν ένα σωρό α, πιθανότητες. Παρακαλώ να το ελέγξετε. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, όλοι έθεσαν δύο ερωτήσεις. Ε, δεν μου απαντήσατε. Είστε μόνος άνθρωπος στον κόσμο που πιστεύετε ότι ο κύριος Μέρτσι ε, δεν είναι ε, ένοχος. Για την Transparency International μπορείτε να μου πείτε τα σχόλιά σας για το, όσα είπε ε, η οργάνωση αυτή ότι η Μάλτα δηλαδή είναι μια από τις πιο διεφθαρμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ απαντήστε μου. Ευχαριστώ. Αναλύς Ντότς. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω παρακολουθήσει ολόκληρη την ακρόαση, αλλά την παρακολουθούσα από το διαδίκτυο και έχω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δικές σας ιδιότητες. οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος, τέταρτη εκδοχή. Ε, Κτιμώ το αυτό που είπατε ότι θα εξασφαλίσετε την επιτυχία. Θέλω να σας ρωτήσω για την θέση του, της Κομισιόν ότι θα πρέπει να καλύπτονται και τα καταπιστεύματα από εδώ και στο εξή σε αυτό τα μητρώα διαφάνειας. Πώς θα το κάνετε αυτό, μήπως είναι πολύ στενός ορισμός και πολύ ε, πολλά τέτοια καταπιστεύματα που θα έπρεπε να, κατα... να περιλαμβάνονται δεν θα περιλαμβάνονται. 2011, έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας λέει ότι υπάρχουν τεράστια εμπόδια στις έρευνες ε, και ότι πολλές φορές είναι τόσο περίπλοκοι αυτοί οι οργανισμοί που είναι δύσκολο να ε, τους ελέγξει κανείς. Ε, πολύ επικίνδυνο αυτό. Πώς θα τα καταφέρετε εσείς και για το Brexit. Ε, ίσως θα μπορούσατε να πείτε ότι θα προσπαθήσετε να επιβάλλετε την ψυχραιμία. Πολύ το χαίρομαι που το είπατε αυτό. Καμιά φορά πιστεύω και εγώ στη χώρα μου ότι κάποιος πρέπει να μας λούσει με κρύο νερό για να συνέλθουμε στη χώρα μου. Πάντως υπάρχουν διάφορα ρυθμιστικά θέματα όσον αφορά το CNU ε, δεν έχουμε πρόβλημα γιατί προφανώς δεν έχουμε ε, ομαλά λειτουργούς, ε, λειτουργών σύστημα για τις αντιστοιχίες, ας πούμε για την τιτλοποίηση. Πιστεύετε πως μια προσέγγιση omnibus ή κάτι αντίστοιχο θα είναι απαραίτητο. Ας ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Όταν γίνει αξιολόγηση του FSP που γίνεται κάθε πέντε χρόνια και νομίζω θα γίνει κατά το δεύτερο μισή του χρόνου μια αξιολόγηση του συνολικού συστήματος στη Μάλτα. Το θέμα είναι ότι οι αρχές, οι φορολογικές αρχές, η αστυνομία θα έχουν πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο. παρόλο που δεν υπάρχει διαφάνεια για το κοινό. Αυτή είναι η φύση του συστήματός μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δεν αποκρύπτονται από τις ε, αρμόδιες αρχές, τις αρχές ε, κατά του ξεπλήματος χρήματος, τις φορολογικές αρχές και την αστυνομία. Αυτό ισχύει, μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Το θέμα ε, της δημοσιοποίησης λοιπόν είναι ε, κατά πόσο είναι προσβάσιμα στις αρμόδιες αρχές ή στο κοινό, συμπεριλαμβάνοντας και τα ΜΜΕ. Έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά θέλω να σταματήσω εδώ. Ας πάρουμε τα έγγραφα του Παναμά, ε, δημοσιοποιήθηκαν και οι εθνικές μας αρχές ε, ξεκίνησαν να εργάζονται με τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους δεν μπορούσαν να πάρουν ούτε από το ICIJ ή από τις αρχές του Παναμά τα στοιχεία αυτά. Άρα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Γι' αυτό ε, προσυπογράψαμε όλες τις συμφωνίες για την ανταλλαγή στοιχείων και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τον ΟΣΑ, γιατί ακριβώς έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα, ε, παγκόσμια εμβέλεια ούτε ώστε βαθμία και βαθμία περιλαμβάνει όλες τις χώρες. Ε, θέλουμε και τους άλλους να συνεργαστούν μαζί μας, δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είναι σημαντικός ο ΩΣΑ, όπως σας είπα. Τώρα, όσον αφορά το Brexit, νομίζω ότι σας ε, γνωστοποίησα τις απόψεις μου. Βεβαίως πιστεύω ότι και δύο πλευρές θα υποφέρουν. Εφόσον υπάρχει, υπάρχουν κάποιες ε, υπηρεσίες, ε, υπάρχει μια αμοιβαία κοινωνία η οποία θα μπλοκαριστεί θα υπάρξει κατάθμιση κλπ. Αλλά δεν θα ήθελα να διατυπώσω εικασίες σε σχέση με το τι θα συμφωνηθεί. Αλλά ευχόμαστε, ευχόμαστε το μικρότερο κακό και για τις δύο πλευρές, το οποίο θα μπορέσει να γίνει αποδεκτό και από τους δύο και πάλι. Ευχαριστούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τη διαδικασία κάτσε γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Υπουργό κύριο Τσικλούνα για αυτή την εξαιρετικά γόνιμη και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Ε, σας εύχομαι τα καλύτερα για την θητεία σας θα ήθελα να εξασφαλίσουμε αμοιβαία την συνεργασία μας. Αναφέρατε και την δέσμευσή σας να προχωρήσετε στο τομέα της φορολόγησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τι συνάδελφοι, θα περάσουμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης στη λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ε, η αρμόδια της Επιτροπή είναι ΙΜΚΟ, συντάκτης ε, γνωμοδότησης τόρου, τόρου Κλαουδιαν Φραντσούλητσα, θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για να ξεκινήσω θα ήθελα να υπογραμμίζω, να υπογραμμίσω ότι έστω και αν η δικαιόχρηση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της ε, κοινή αγοράς, και στο λιανικό εμπόριο δεν έχει πετύχει το δυναμικό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μιας κακής εφαρμογής του κανονισμού. Η έλλειψη ομοιογένεια στην εφαρμογή του σε όλα τα κράτη-μέλη υπονομεύει την αποτελεσματικότητα του κανονισμού 330-2010 της Επιτροπής και θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη να αναθεωρηθούν οι διατάξεις για την εφαρμογή του κανονισμού από τις χώρες μέλη. Η υλοποίηση του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο και η εφαρμογή του θα πρέπει να προσαρμοστεί ούτω ώστε να επιτύχει πιο αποτελεσματικά τους στόχους. Έχουμε, θα πρέπει να διατυπωθεί καλύτερα το κανονιστικό πλαίσιο των ε, συμβάσεων ε, ε, franchising, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αμεροληψία. Είναι σημαντικό να δούμε τον κανονισμό και να τον αναθεωρήσουμε και γι' αυτό θα πρέπει να επεληθεύσουμε τις επιπτώσεις της οριζόντιας στρατηγικής σε σχέση με την λειτουργία της δικαιόχρησης. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις και την αναλογικότητα των ε, κάθετων ε, περιορισμών. Ε, θα πρέπει να έχουμε εμπορικά πληροφορίες για τις νέες τάσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να προσαρμόσουμε το κανονισμό στην ψηφιοποίηση της οικονομίας. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι για να απλωστεύσουμε τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών για την κατάσταση στην αγορά, ένα μοντέλο δήλωσης ή κοινοποίηση θα πρέπει να δημιουργηθεί. Μία περιεκτική ανάλυση των ε, διαφορών που υπάρχουν ε, στις εθνικές αγορές θα μπορούσε να υπάρξει δημιουργώντας πληροφορίες για ε, περιπτώσεις ε, χρεοκοπίας, πτώχευσης. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την, ε, να εντοπίσουμε τα αθέμητα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχουν ορισμένες χώρες μέλη και να να εκκινήσουν οι αναγκαίες διαδικασίες έρευνας. Ελπίζουμε ότι ο κανονισμός θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2018 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει ενεργά στην προσαρμογή του κανονισμού και τις ε, οδηγίες για τη δικαιόχρηση. Η δικαιόχρηση είναι ένα σημαντικό θέμα για την οικονομία της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για εκ μέρους του ΕΛΚ, ο Ιγκογκάρ Πέλτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε, καθώς και τον πρώτο αντιπρόεδρο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στα επόμενα δυόμιση χρόνια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φρονζούλικα για το κείμενο της ε, γνωμοδότησής του. Νομίζω ότι περιέχει πολύ καλές προτάσεις. Ο εισηγητής ε, πολύ καλά έχει περιγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα αυτών. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις προτάσεις. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστά αιτιολογημένες. Έχω τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλλω. Πάντως νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά πάνω στο θέμα αυτό. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να εξαλείψουμε τα προσκόμματα για την καλή λειτουργία της ενίας αγοράς. Υπάρχουν όμως ε, και κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να τηρούνται. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι επί της ουσίας αρμόδια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με τα θέματα που εμπίπτουν στις δικές μας αρμοδιότητες, ε, κυρίως δηλαδή ε, το δίκαιο περί ανταγωνισμού. Ε, ο κύριος Φρουνζούλικα ασχολείται εδώ και με αθέμητες πρακτικές. Δεν υπάρχουν, ε, δεν αρκεί εδώ το κανονιστικό πλαίσιο. Στο σημείο 16... Η πρόταση κειμένου αναφέρεται στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε σωστό κανονιστικό πλαίσιο, δεν είναι όμως σαφές το αν χρειαζόμαστε συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή αν χρειαζόμαστε νομική πράξη. Όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, μας περιμένει πολλή δουλειά νομίζω. Όπως αναφέρεται και στο κείμενο, οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ιδιαίτερα στις συμβάσεις B2B. Χρειαζόμαστε λοιπόν σχετικά μέτρα και θα υποβάλουμε σχετικές τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι χρέος μας στην νομοθεσία να υπάρχει επαρκής ασφάλεια στο θέμα αυτό. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά. Και συμφωνώ και με τη δομή που έχει δώσει ο συντάκτης ε, στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιον από το ECR, όχι. Ούτμαν Κρέσπο, όχι. Υπάρχει κανείς που θέλει να πάρει το λόγο από άλλη ομάδα, εάν όχι, να δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που δεν είναι παρόντες άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάντως ε, την Ουγγαρέζα συνάδελφο. Πάντα εκτιμώ τις παρεμβάσεις της. Φυσικά θα συνεργαστούμε. και ο τελικός στόχος είναι να συμβάλλουμε στην αλλαγή των κανόνων μέχρι το τέλος του 2018 στο θέμα της δικαιόχρησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. 8 Φεβρουαρίου προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, 9 Μαρτίου εξέταση των τροπολογιών. Ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ 27 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτουσίας Αρμόδια Επιτροπή 25 Απριλίου. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση του κανονισμού 99-2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα με παράτασή του για την περίοδο 2018-2020. Είμαι εγώ εισηγητής. Η ανάγκη για στατιστικά στοιχεία αυξάνεται, όπως όλοι γνωρίζουμε. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με συγκεκριμένες αρχές και γι' αυτό έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πέρσι τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επίτροπη υιοθέτησε πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού 99-2013 για το στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017 ε, για την παράτασή του για την περίοδο 2018-2020. Αναγνωρίζω ότι τα εθνικά στατιστικά συστήματα ε, έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για εξυγχρονισμό ε, του τρόπου λειτουργίας τους. Ωστόσο, πρέπει να καλυφθούν κάποια κενά, ώστε οι στατιστικές να μπορούν να στηρίζουν τις διάφορες πολιτικές ιδιαίτερα τις ε, πολιτικές προτεραιότητες ε, της Κομισιόν. Γενικά, στηρίζω την πρόταση της Επιτροπής, ε, που στόχο έχει να βελτιώσει την συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, έχω υποβάλει 18 τροπολογίες για να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία που λείπουν από την πρόταση. Σε τέσσερις ιδιαίτερα τομείς προτείνω τροποποίηση. Καταρχάς, να να λάβουμε υπόψη την κατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ε, συμφωνώ με την ανάπτυξη μεθοδολογίας ε, για έρευνα, για την ε, βία με βάση το φύλλο. Τρίτον, κοινή νομική βάση για κοινωνικές στατιστικές και τη δημιουργία κοινή υποδομής και κοινών εργαλείων. Τέταρτον, ενθαρρύνω την ανάπτυξη για τρόπους ε, εξέτασης ε, των διαφόρων μορφών απασχόλησης, μερικής ολικής, ε, περιορισμένου χρόνου κλπ. Πέμπτον, να εξετάσουμε την περίπτωση πιθανής αποχώρησης από την Ένωση μέλους, κράτους μέλους. Και τέλος, τροπολογία όπου ζητώ άμεσα έκθεση και μια οριστική έκθεση που θα εξετάζει την ε, αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων. Επικροτώ την γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, διότι γενικά ευθυγραμμίζεται με την ε, προσέγγιση που προτείνω εγώ και περιμένω να ακούσω τις παρατηρήσεις σας και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να εξετάσουμε πιθανές τροπολογίες. Από το ΕΛΚ και εκ μέρους του κυρίου Μάτο, ο κύριος Κάρλος Ιτουρκάκης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο στο όνομα του κυρίου Μάτο που δεν μπορούσε να παρακολουθεί στη σημερινή συνεδρίαση γιατί έπρεπε να βρίσκεται σε άλλη ε, επιτροπή αυτή τη στιγμή. Ε, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν εξ ονοματός του καταρχάς τον εισηγητή και τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, που ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Η Κομισιόν παρουσίασε τις πολιτικές προτεραιότητες και τη σημασία να ανταποκριθούμε στην ολοένα και ξενόμενη ζήτηση για στατιστικές και την ταχύτερη εκπόνησή τους και γι' αυτό η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών θα πρέπει να βασίζονται σε συγκρίσιμες στατιστικές και υψηλής ποιότητας για την οικονομική, την περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση στην Ένωση, καθώς και στις συνιστώσεις τους σε κλίμακα εθνική ε, και για τις περιόδους 18 με 20, να εξασφαλίσουμε ότι θα καλύψουμε τρεις ε, στόχους βασικούς, που πρώτος είναι η ενημέρωση και οι στατιστικές υψηλής ποιότητας, να μην υπάρχουν ελλείψεις στις στατιστικές. Δεύτερον, να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα στις ανάγκες τις στατιστικές της Ένωσης και τρίτον να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και κατά αυτόν τον τρόπο να εγγυηθούμε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό ο κ. Μάτο μου είπε ότι παραμένει στην διάθεσή σας, Πρόεδρε, ώστε να εγγυηθούμε την ολοκλήρωση αυτών των στόχων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβες που είναι. Ε, σκιώδης εισηγητής, ε, τώρα για την ΚΟΕ, ο κύριος Βιέγας. Έχετε το λόγο, μάλιστα πολύ σύντομα. Εμείς εν Συμφωνούμε με το περιεχόμενο της έκθεσης. Όντως ε, πρόκειται για βασικά εργαλείο για να μπορούμε να αναφερόμαστε στο και να μετράμε την ορθότητα των στατιστικών και των πολιτικών που ασκούμε κατά συνέπεια. Ε, με, πρέπει όντως να είναι καλής ποιότητας. Ε, είναι σωστό να τελειοποιηθούν κάποιε πτυχές των στατιστικών που έχουν να κάνουν με κοινωνικά και εργασιακά θέματα. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη να απομαδοποιηθούν οι ε, συμβάσεις αορίστου χρόνου και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επίσης, είναι σημαντικό να καταγράφονται οι μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες, τα θέματα του φύλου, τα θέματα των μεταναστών και ούτε καθεξής. Επίσης, θα μπορούσαμε εδώ να ξεκινήσουμε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη και που σχετίζονται με φορολογικά ζητήματα. Είναι ε, τα θέματα που μπορούν να μας βοηθήσουν ε, να αντιμετωπίσουμε τα, τα οικονομικά ζητήματα, το tax gap, τα διάφορα που δυστυχώς υπάρχουν ε, και που υπάρχουν κάποιοι σύνθετοι δείχτες αυτή τη στιγμή που στην ουσία επιτρέπουν ε, το να εκπονούνται αξιόπιστες στατιστικές. Και αυτό θα δούμε πώ θα μπορέσουμε τώρα να τα θέσουμε όλα αυτά σε εφαρμογή. πάντω. Ε, για την ώρα είναι θετικό ε, το μήνυμα και συμφωνούμε με τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους ορτασούν. Μάλιστα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να, να δούμε ε, με συγκεκριμένα σημεία. Καλωσορίζουμε την έμφαση που δίνει ο εισηγητής σε ευρύτερα στατιστικά στοιχεία για να ορίσουμε τι κοινωνικέ στατιστικές αλλά και να δούμε το εξελισσόμενο τοπίο για τις μεταναστευτικές ροές. Αυτά ε, συνάδουν με την ε, ατζέντα για την ανάπτυξη. Τα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μετρήσουμε και τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό είναι δύσκολο, ωστόσο λείπουν και κάποια στοιχεία, ε, γιατί η Eurostat έχει μείνει πίσω σε σχέση με την στατιστική εργασία το ΟΗΕ σε αυτό το τομέα. Όπως αποκαλύπτεται από το site της ε, Eurostat, βασικοί δείκτες της στρατηγικής για το 2020 ε, λείπουν γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, πούμε, για τις εκπομπές ε, ρίων του θερμοκηπίου ε, λέει για την ενέργεια και την κατανάλωση της πρωτογενούς και της τελικής ενέργειας. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως αφορούν το 2014. Παρότι είχαμε διάφορες ανταλλαγές απόψε με εκπροσώπους της Eurostar για το πώς θα βελτιωθεί η πρόσβαση στα στατιστικά του στοιχεία, η ανάκτηση και η εφαρμογή των στόχων της Eurostat και των πόρων της Eurostat φαίνεται να είναι επιβαρυντική για τον απλό πολίτη. Ε, μετά από τροπολογία που έχει κατατεθεί. Θα πρέπει να βελτιωθούν ε, τα στοιχεία, όπως είπαμε, για το στόχο του 2020, τα κοινωνικά και τα θέματα αλληλεγγύης και επίσης να βελτιωθεί η, ε, δυνατότητα χρήσης ε, για τους απόλυτες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τον εισηγητή για την πρότασή του. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Σιώδης για την ε, επικοδομική τους συμβολή και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μια πολύ καλή συνεργασία που θα καταλήξει σε ένα καλό κείμενο και σύντομα θα ξεκινήσει το τριμερείς συναντήσει. Η προθεσμία για τι τροπολογίε 8 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, η εξέταση τροπολογιών στις 9 Μαρτίου, 27 Μαρτίου στην ΙΜΚΟ η ψηφοφορία, στην Ολομέλεια στη σύνοδο του Ιουνίου του 2017. Αλλά δική μου πρόθεση είναι να συνεχίσουν άμεσα οι τριμερείς ε, συνεδριάσεις. Ωραία, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ε, βλέπω ότι οι ομάδες διανέμουν ακόμα τους καταλόγους, τις λίστες ψηφοφοριών. Θα περιμένουμε λίγα λεφτά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 Συγγνώμη, Πρόεδρε, για σήμερα είναι η ψηφοφορία ή άλλη μέρα. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Και υποτίθεται θα ξεκινούσαμε 11 και 10. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Καταρχάς μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Σας παρακαλώ καθίστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Colleagues, please vote. Συνάδελφοι, παρακαλώ ψηφίστε. Can I have it closer? I would like to see it. Still some six colleagues have put a card but they are not voting. I encourage all... Εξή συνάδελφοι έχουν τοποθετήσει την κάρτα τους ε, αλλά δεν έχουν ψηφίσει όλοι. Παρακαλώ. And one still colleague to vote. Ελέγχουμε και τη σύνθεση. Ένας ακόμα απομένει να ψηφίσει, σας παρακαλώ. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο θέμα. Είναι το προσπέκτου στο ενημερωτικό δελτίο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Γέζεκ. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω τον ε, προκάτοχό μου, τον Φιλίπ Τεπάκερ, που ξεκίνησε τη διαδικασία εδώ στο Κοινοβούλιο και να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές. Διότι ήταν συνεργάσιμοι και επικοδομητικοί περισσότερο από ποτέ. Έτσι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Το οποίο κάνει τη χρηματοδότηση λιγότερο δαπανηρή και πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ και την Γραμματεία, τον Πρόεδρο και άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Έναρξη της ψηφοφορίας. Technical problems. We start again. Έχουμε τεχνικά προβλήματα. Ξεκινάμε πάλι. Παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας 44 υπέρ, 8 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια. Προχωράμε στην έκθεση του Φίλιπ Λάμπερτ. Είναι πολύ μακρύς ο τίτλος, δεν θα τον διαβάσω λοιπόν. Και θα ψηφίσουμε μαζί τις ε, τροπολογίες 10 και 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την συμβιβαστική χωρίς την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C με προφορική τροπολογία. Έχω αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Παρακαλώ λοιπόν όσοι συμφωνούν μαζί μου να το δείξουν. Τέσσερις βλέπω. Συμβαστική C χωρίς ε, την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 4 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 50 δεν είναι παραδεκτή. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική e, ε. Αλλά μέχρι το set out in article 2 διότι το τελευταίο τμήμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΙΜΚΟ, σύμφωνα με την κοινή συμφωνία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία, αυτά 10 παράγραφος 1 του εισηγητή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 ΙΜΚΟ υπέρ κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. ΙΜΚΟ 4. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση Ήμκο 8. Παρακαλώ. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 23 υπέρ. Α, καταπίπτει. 24. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Απορρίπτεται. Συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος, λέει ο πρόεδρος. Λάθος έκανα, απορρίπτεται σαφώς. 25. Υπέρ κατά αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 25. Is adopted εγκρίνεται κατά δύο ψήφους. Η 9 καταπίπτει, όχι, είναι συμβατή, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 12, υπέρ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση, ΙΜΚΟ 12, παρακαλώ. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. 31, δεν βλέπω τα χέρια σας. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Still two colleagues to vote. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Α, ε, νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί ε, τις 6, 7, 8 και 9 τις επιλογές αναφορές υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Ονομαστική ψηφοφορία πάνω στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Αρχή της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Ονομαστική ψηφοφορία πάνω στο νομοθετικό ψήφισμα. Υπέρ. Λήξη της ψηφοφορίας. 49 υπέρ, 2 ε, κατά 5 αποχές. Ε, ψηφοφορία πάνω στην απόφαση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έναξη της ψηφοφορίας. Is adopted. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. εγκρίθηκε η εντολή, καθώς και η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Ε, ε, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, εισηγητής, εσκιώδης ε, και εισηγητής της ΙΜΚΟ. Έχουμε λοιπόν αυτήν την νέα διαδικασία. Πρόκειται για την απόφαση που λάβαμε για την ένταξη των διαπραγματεύσεων που θα ανακοινωθεί στο, κατά την ένταξη της Συνόδου και μέχρι το τέλος ε, αυτής της ημέρας, ε, μέχρι το 1 δέκατο των ευρωβουλευτών, τουλάχιστον το 1 δέκατο των βουλευτών μπορεί να ζητήσουν ε, ψηφοφορία πάνω στην απόφαση αυτή και στην περίπτωση αυτή το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει κατά τη διάρκεια της ίδιας περίοδου νόδου. Αλλιώ θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Προχωράμε τώρα στο σχέδιο έκθεση τη Ντανούτα Χούπνερ. Ε, για την Τραπεζική Ένωση. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 88. Η 88 είναι... Very strange, but so amendments 88 and 110. 88 και 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το ελέγξουμε έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε πρώτα τη συμβιβαστική C σε συμφωνία με την εισηγητρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι, e, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 174 έναξη ψηφοφορίας. Vote Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 183 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 183 ένευση ψηφοφορίας. Vote Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική J υπέρ κατά... Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε τώρα στην προφορική τροπολογία πάνω στην παράγραφο 7α των πρασίνων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά... Νομίζω ότι απορρίπτεται η ηλεκτρονική επαλήθευση ε, έναξη ψηφοφορία. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική J α υπερκατά κατά αποχές εγκρίνεται, 2.46 υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική Κ. υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική Λ υπέρ αποχές εγκρίνεται. 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία των πρασίνων πάνω στην παράγραφο 8α υπέρ. Κατά. Α, νομίζω ότι εγκρίνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση έναξης ψηφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική M. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.41 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 2.41 τη ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 2.47 έναρξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Yes, was. Compromise MA in... Συμβαστική MA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική MB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία των πρασίνων για την παράγραφο 9 γ υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, η ένταξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο. 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 269 Έναξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 272 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 272 Έναξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 2,73 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 2,74 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Όπως και πριν θα ψηφίσουμε πρώτα τη συμβαστική νη. Εν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2,76 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 289 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 288 και 240 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 307 υπέρ. Συγγνώμη, 307 καταπίπτει. 275 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Ω όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική π, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία των πρασίνων πάνω στην παράγραφο 12α υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση έναξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 311 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.32 και 3.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Still three colleagues to vote. No? Yes? Okay. Let's close the vote. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16α, προφορική τροπολογία των πρασίνων. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική U, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική V. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Όχι. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. Δι, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική W, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 356, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 255, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική WA υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AC υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. 4.15 υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. 4.16 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 416 έναρξη ψηφοφορία. Vote is Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 4.35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.36 υπέρ. Τι ψηφίζει το ΕΛΚ στο 4.36 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση 4.36 έναξης ψηφοφορίας. Vote is closed. Is Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 4.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. Τροπολογία 1 υπέρ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 το αρχικό κείμενο. Οι 7 καταπίπτει. Έχουμε το αρχικό κείμενο. Ε, αιτιολογικές αναφορές 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 8 και 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, αιτιολογική αναφορά 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, το αρχικό κείμενο, ε, ε, αιτιολογική αναφορά 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ψηφίζουμε μαζί από την 11 έως την 25. Από την 11 στην 20. Συμφωνείτε? συμπεριλαμβανομένου του αρχικού κειμένου στο σημείο 6 έως 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 21 υπέρ. 21. Exactly. Don't need to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 Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, είχαμε ζητήσει να ψηφίσουμε μαζί μέχρι την 17. Έστω και την αιτιολογική αναφορά 14, το αρχικό κείμενο. Θα χάσουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι θα κερδίσουμε. Δεν ήταν λοιπόν πολύ καλή η απόφαση αυτή. Διότι ψηφίζουμε πράγματα που αντιφάσκουν μεταξύ τους. Η 11 κάνει να καταπέσει η 13. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό λοιπόν. Uh, Μία-μία θα τις ψηφίσουμε, διότι αλλιώς δεν είναι σαφές τι ακριβώς γίνεται. 11 υπέρ. Καλή απόπειρα κύριοι συντονιστές, αλλά 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 καταπίπτει, 12 υπέρ εγκρίνεται, 14 υπέρ εγκρίνεται, 15 υπερ αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο ε, Αιτιολογικές αναφορές 10-13 υπέρ εγκρίνεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 17 καταπίπτει. Αρχικό κείμενο, αιτιολογική αναφορά 14 υπέρ κατά εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά εγκρίνεται, αρχικό κείμενο αιτιολογικές αναφορές 15, 20 υπέρ αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο 21 υπέρ κατά εγκρίνεται, 21, τροπολογία 21 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 21, έναξης ψηφοφορίας. bodies. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο και αναφορά 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 κατά 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, αιτιολογικές αναφορές 23-25, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπερκατά κατά αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο, αιτιολογική αναφορά 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική αναφορά 27, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του 28, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 27, έναρξη της ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της αιτιολογικής αναφορής 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 30 υπέρ κατά τα... Α... Τι ψηφίζει το ΕΛΚ υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική AD υπερκατα κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 79 έναρξης ψηφοφορίας. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση της 46 έναρξη ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Κατά μία ψήφο 48 υπέρ. Κατά 48 ηλεκτρονική επαλήθευση έναρξη ψηφοφορίας. is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, έναρξη της ψηφορίας. 64. Λήξη της ψηφοφορίας. Ισοψηφία. 26 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. Τροπολογία 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση έναξη ψηφοφορία. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Okay, I can. Is 66. 66, τροπολογία 66, έναρξη της ψηφοφορίας. Still one colleague to vote. Before he had voted. Now not. I Okay. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά ποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62, 72, συγγνώμη, διορθώνει ο Πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση της 80. Vote is closed. Is rejected. Απορρίπτεται. There was 80, so 81. Ψηφίσαμε την 80 λοιπόν, 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφοφορία πάνω στο κείμενο όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 45 υπέρ, 11 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Now I have to announce that uh, the joint Econ Badge... Η κοινή συνεδρίαση Econ Badge, η ψηφοφορία ε, έχει αναβληθεί οι εισηγητές θα υποβάλουν την έκθεση κατά την δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το τμήμα της συνεδρίασης. Θα συνεχίσουμε στις 3. Ευχαριστώ.